Στι 11 Ιανουαρίου έλαβα μια επιστολή από τους Πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων και Πρασίνων όσον αφορά τη συμπεριφορά των υπρόεδρων τσαρνέστ και ζητείται η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 21 του κανονισμού του Κοινοβουλίου στη συνέχεια κάποιων δηλώσεων άλλου βουλευτού στο Ευρωκοινοβούλιο. Το θέμα συζητήθηκε από την διάσκεψη των πρόεδρων σε δύο διαδοχικές ε, ε, συνεδριάσεις 18 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου. Στις 18 Ιανουαρίου επίσης το επιστολή του Αντιπρόεδρου Τσαρνέσκη όπου απαντούσε σε αυτά τα οποία αναφέρονται στην προηγουμένη επιστολή. Στις 23 Ιανουαρίου ε, είχαμε την ακρόαση του κυρίου Τσαρνέσκη για το θέμα και λήφθησαν υπόψη τα όσα είπε στις 1η ε, Φεβρουαρίου αποφάσεις ιδιαίτερα των Προέδρων με μία πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψήφισάντων να, και επί τη βάση τριών πολιτικών ομάδων να προτείνει το πέρας της εντολής του Αντιπρόεδρου δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο την ε, Τετάρτη πρόκειται να αποφασίσει και απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων και πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το σώμα αυτό. Έχετε το λόγο. Σε... Διαδικαστικό. Teraz, panie przewodniczący, w związku z tym Έχω μία ερώτηση, Πρόεδρε, σε σχέση με το εξή ζήτημα. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα μόλις είπατε, η ερώτησή μου είναι η εξής. Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λογοκρίνει από εδώ και πέρα ε, τις δηλώσεις των Ευρωβουλευτών στα κράτη-μέλη τους. Δεύτερη ερώτηση. Πότε θα αντιδράσει το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στις σκανδαλώδεις δηλώσεις του κυρίου Φερχόφστατ ε, που προσέβαλε την, ε, το πολωνικό έθνος εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Κάτι πρωτοφανές. Θα τιμωρήσετε λοιπόν αυτά που λένε οι ευρωβουλευτές εκτός του ημικυκλίου με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Το άρθρο 21 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, λέει ο πρόεδρο ορίζει ότι τότε μόνο προέρχεται από τρει κοινοβουλευτικέ ομάδε που έχουν εκπροσωπούν την πλειοψηφία και δεν πρόκειται για κάποια κύρωση του κανονισμού που επιβάλλεται che Επιβάλλεται από τον πρόεδρο, ούτε απόκειται στον πρόεδρο, ούτε απόκειται στο Προεδρείο να αποφασίσει. Αυτοί οι οποίοι κρίνουν είναι τα μέλη τη διασκέψεω των Προέδρων. Επομένω, πρόκειται για αίτημα των κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν είναι κύρωση με αυτή την έννοια. Πρόκειται για εφαρμογή Βάρτρο 21. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να εφαρμόσω τον κανονισμό. Εάν αυτό κρίθηκε με ψηφοφορία στην διάσκεψη των ε, πρόεδρων, αυτό σημαίνει ότι τηρήθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία. Δεν πρόκειται για κάποιε κυρώσει από πλευρά του πρόεδρου. Δεν μπορεί ο πρόεδρο να επιβάλλει κυρώσει για κάτι το οποίο συνέβη εκτό κοινοβουλίου. Μόνο για ό,τι συμβαίνει εδώ, στο κοινοβούλιο. Το αίτημα του να παυθεί από τα καθημερινά του ως αντιπροέδρου είναι κάτι το οποίο το ορίζει το άρθρο 21 ετήσιο κοινοβουλευτικών ομάδων, πολιτικών ομάδων. Κύριε Βέμπερ, έχετε το λόγο. Η συνάδελφος κύριε Πρόεδρε μιλάει για την ελεύθερη έκφραση και δεν περιορίζεται η ελεύθερη έκφραση Περιμένουμε από εσά, κύριε Πρόεδρε, να κρατήσετε μια ουδέτερη θέση και το κάνετε εσεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, όπω περιμένουμε και από του άλλου αντιπροέδρου να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, όπω αρμόζει σε ένα όργανο όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όταν έχουμε έναν αντιπρόεδρο, ο οποίο ε, ε, περιγράφει ε, κάποιους ως ναζί που ε, περιγράφει ε, ε, κάποιους με τη Σοβιετική Ένωση ίσως να έχουν περαστεί κάποιες κόκκινες γραμμές. Mm. και η ομάδα μου είναι έτοιμη να ε, σκεφτεί κάποιον άλλο εκπρόσωπο ως αντιπρόεδρο γιατί δεν πρόκειται για θέματα Πολωνίας ή για θέματα πολιτικής ομάδας. Εμείς είμαστε υπέρ οποιοδήποτε άλλου συναδέλφου τον οποίον θα προτείνει το ECR αλλά για το συγκεκριμένο συνάδελφο νομίζω ότι θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Ο κύριο Μπούλμαν έχει το λόγο, αλλά να μην συζητήσουμε τώρα για τον κύριο Τσανέσκη, διότι η απόφαση έχει ληφθεί. Πρόκειται να γίνει ψηφοφορία με, ε, με τρόπο μυστική ψηφοφορία και αδώ το λόγο στον κύριο Μπούλμαν. Αλλά ε, απλώ από πλευρά ε, νομική απάντησα προηγουμένω, γιατί αναφέρθηκε ε, στο οποίο επέβαλε την, ε, την κύρωση ο πρόεδρος ή το προεδρείο. Όχι, ήταν κάτι το οποίο ε, επευλήθη ως κύρωση από το άρθρο 21. Είναι κάτι το οποίο περιβάλλεται από τις σχετικές εγγυήσεις ακόμη και να επρεστεί τον αυτός ο κύριος Τσάρνες και σας είπα τι έγινε. Οπότε όλα έγιναν όπως προβλέπεται. Κύριε Μπούλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ούτε και εγώ θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση από αυτού. Άκουσα την ερώτηση της συναδέλφου και θέλω να απαντήσω. Όχι, στη διάσκεψη των Προέδρων ε, δεν ε, ακούστηκε τίποτα για ε, λογοκρισία. Ούτε θα γινόταν κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ενότητα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της άρνησης του εθνικοσοσιαλισμού και του πολέμου και οποιοδήποτε χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις ξεπερνάει πραγματικά μια κόκκινη γραμμή και οι σοσιαλδημοκράτες, η δική μας πολιτική ομάδα δεν θέλει να εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κάποιον ο οποίος κάνει τέτοιες συγκρίσεις ε, με ναζί. Ούτε ναζί ε, έχουν θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τέτοιες δηλώσεις και είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε. Εξάλλου, συμφωνούμε με τον συνάδελφο Βέμπερ και είμαστε κι εμείς ε, έτοιμοι να εκλέξουμε ένα εκπρόσωπο ή μία εκπρόσωπο που δεν θα ξεπερνάει αυτά τα όρια. Είμαστε υπέρ της ε, πολυμορφίας ε, και της ε, διαφορετικότητας στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν δεχόμαστε κανένα ναζί και κανέναν εκπρόσωπο των ναζί. Λάμπερτ, σας ξαναλέω, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα συζήτηση. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θέλω να στηρίξω τη δική σας θέση, Πρόεδρε. Πολύ σωστά το χειρίζεστε. Εγώ εδώ σε αυτό το ημικύκλιο είμαι υπέρ των αντιμαχόμενων επιχειρημάτων ε, αλλά άλλο αυτό και άλλο η προσωπική προσβολή όπως αυτήν την οποία προέβη ο κ. Τσαρνέσκι. Ε, όλοι έχουν το δικαίωμα σεβασμού, όλοι μας έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και ο κύριος Τσαρνέτσκι ε, δεν ε, τήρησε αυτή την αρχή. Ευχαριστώ. Κύριε Φορέντζο, και εγώ πρώτα θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να ε, γίνει αυτή η διαδικασία για την οποία ε, ως επιστολή υπάρξαν πάνω από 100 συνάδελφοι δεν είναι δυνατόν να έχουμε πρόσβαση στο κοινοβούλιο τέτοιων ε, πολιτικών δυνάμεων όπως το Casa Pound που είναι οι φασίστες του 21ου αιώνα. Είδατε τι έγινε στην ε, Ματσεράτα. Θα πρέπει μενώς όλα αυτά να τα καταστήλουμε με αποφασιστικότητα. Κυρία Φορέντσα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που διέπουν τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επιτρέψει ή να απαγορεύσει κάποιες πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Ε, όμως, όταν έχουμε τέτοιες ε, τοποθετήσεις, εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω σε έναν βουλευτή εκτός μικροφώνου. Δεν ωφελεί να φωνάζετε. Καθίστε και σεβαστείτε την σειρά σας. Πολύ καλά. Έτσι είναι η δημοκρατία. Συνεχίζει εκτός μικροφώνου ο βουλευτής. Δεν ωφελεί αυτό το οποίο κάνετε. Δεν έχετε ζητήσει το λόγο. Ηρεμήστε ούτως ώστε την υφάλεια να τοποθετηθούμε πολιτικά. Σας ανακαλώ στην ε, τάξη και στην ευγένεια. Πρόεδρος, όταν κάποιος πρέπει να τοποθετηθεί και όταν έχουμε ε, παραβίαση του δικαίου δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τίποτε άλλο. Αυτό ακριβώς ε, και εμείς τώρα κάνουμε όσον αφορά την εκδήλωση για, την, ε, για το στην ε, Ματσαράτα. Δεν είναι θέμα ε, του να επιτρέψουμε ή να απαγορεύσουμε. Είναι θέμα του τι γίνεται μέσα στο Κοινοβούλιο και τι όχι. Όλοι οι βουλευτές είναι ίσοι. Ποτέ έχουμε όμως κάποιες δηλώσεις που παραβιάζουν τον κανονισμό δεν μπορούμε παρά να επέμβουμε. Τώρα, στην συνέχεια της ε,